Ο κύριος Δέμες Μάκερ για ένα λεπτό εισηγητής έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι σήμερα 1,2 εκατομμύρια παιδιά περιφέρονται ε, στην Ιγυρία με βαριά ε, ψυχικά τραύματα μετά από τις επιθέσεις ε, των Μπόκο Χαράμ. Πρόκειται για την καταστροφή μια ολόκληρη ε, γενιά. Ο κύριος Μπουχάρη, ο νέος πρόεδρος, πρέπει να προστατεύσει τα παιδιά και σε αυτόν στρέφομαι. Κάντε τη διαφορά γιατί παρά τα πετρελοδολάρια ε, δεν έγιναν προσπάθειες για την προστασία του πληθυσμού είναι στην κορυφή ε, των πετρελοπαγωγών χωρών η Νιγηρία, αλλά ε, στον πάτο σε ό,τι αφορά τι επιδόσει τη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε ε, τη βία, βλέπουμε του αποθαρρυμένου στρατιώτε και βλέπουμε του απλού ανθρώπου να γίνονται θύμα αυτών των των μελών της Μπόκο Χαράμ πρέπει να στείλουμε ένα πάρα πολύ χειρό μήνυμα, όχι μόνο με τα λόγια μας, αλλά και με τις πράξεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Παγάθα Ορτουντούα. You have the floor in minute. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Η Μπόκο Χαράμ είναι το σκληρότερο και πιο αποτρόπαιο πρόσωπο του πολιταρχισμού. Καταστρέφουν ε, την αξιοπρέπεια των κοινωνιών και ακριβώς αυτός είναι ο στόχος τους και γι' αυτό επιτίθεται και κατά των παιδιών που είναι το μέλλον της κοινωνίας. Ε, χρησιμοποιούν ε, το βιασμό, επιτίθενται σε σχολεία. Εμείς όμως πρέπει εκεί που γκρεμίζεται ή επιτίθενται κατά ενό σχολείου να δημιουργούμε ένα νέο σχολείο και να γυρίζουμε πίσω τις γυναίκες που έχουν υποστεί την αξιοπρέπειά τους. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας ε, για την Ιγυρία και έχουμε καταθέσει γι' αυτό το λόγο αυτό το σχετικό ψήφισμα. Δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάμε την Ιγυρία και πόσο μάλλον τα παιδιά. Είναι κάτι που τους το οφείλουμε και το οφείλουμε ως διεθνή κοινότητα. Ευχαριστώ. Ο Κοράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση των παιδιών στην Ιγυρία και οι εκτοπισμοί που οφείλονται στι δραστηριότητε τη Μπόκο Χαράμα στην Ιγυρία είναι σαφέ ότι μα παραπέμπει στη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί σε αυτή τη χώρα που είναι η πιο πλούσια στην Αφρική, μια από τι πιο πλούσιε, αλλά ε, όπου σοβεί και η φτώχεια, ένα παράδοξο και όπου υπάρχουν τέτοιε καταστάσει. Εκατομμύρια παιδιά που ε, εκτοπίζονται, που φεύγουν, ε, που προσπαθούν να ξεφύγουν λείπουν ε, πόροι ακόμα και για το νερό και τα βασικά δικαιώματα για τα παιδιά αυτά. Αυτά με βάση τα όσα μας είπε η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. Θα πρέπει να πιέσουμε τη διεθνή κοινότητα να δώσει τους πόρους αυτούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά είναι παιδιά τα οποία χρησιμοποιούνται και ως στρατιώτες. Ε, και είναι ένα θέμα στο οποίο δεν κάνουμε αρκετά. Υπάρχουν ε, και νέα που φτάνουν και δεν αφορούν μόνο την Ιγυρία και αφορούν αυτό το θέμα των παιδιών στρατιωτών. Θα πρέπει ε, πάντως να κάνουμε κάτι έτσι ώστε όταν φεύγουν από τις παραστρατιωτικές οργανώσεις να μπορούν να ενταχθούν σε συγκεκριμένα προγράμματα. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Παντζέρη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην Ιγυρία η ανασφάλεια που προκαλείται από την ένοπλη σύρεξη μεταξύ της ε, παραστατικής οργάνωσης Μπόκο Χαράμα ε, και των ε, δυνάμεων της τάξης της χώρας έχουν προκαλέσει τον εκτοπισμό πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιών. Δεν υπάρχει πρόβλημα στα τρόφιμα, στο πόσιμο νερό και στις υγειονομικές υπηρεσίες. Τα παιδιά κινδυνεύουν να πεθάνουν από την ελονοσία, την ε, κακή διατροφή και βρίσκονται θύματα μιας ε, ένοπλης σύραξης. Οι νέες γυναίκες έχουν ε, υποστεί αναγκαστικούς γάμους, καταναγκαστική εργασία και ούτω καθεξής. Επίσης τα παιδιά χρησιμοποιούνται και ως ανθρώπινες βόμβες. γι' αυτό και κάνουμε μια έντονη έκκληση να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση από πλευρά της διεθνούς κοινότητας με αρχή, αρχής γινωμένης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η ε, κυρία Χόιμπουκ, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ιγυρία είναι δραματική. Και η Μπόκο Χαράμ έχει συνάψει ε, ανίερη συμμαχία με το Ισλαμικό κράτος. Ε, μία συμμαχία που συνεχίζει να προωθεί την τρομοκρατία στην ε, Ήπειρο αυτή, αλλά και πέρα από την Ήπειρο αυτή. Μόνο αυτό το μήνα έχουν χαθεί 1.600 ζωές ε, από την Ποκοχαράμ και χιλιάδες παιδιά έχουν διωχθεί. Υπάρχουν στην Αιγυρία λοιπόν τόσα πολλά παιδιά που δεν πηγαίνουν στο σχολείο ακριβώς λόγω της τρομοκρατίας ε, της Μποκοχαράμ. Το ανέφεραν αυτό και οι προκαλήσαντες Εδώ η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες της. Και οι υποσχέσεις σε ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια να τηρηθούν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που ο Επιτροπός λοιπόν θα αυξήσει τους, τα κονδύλια για τα θύματα της Μποκοχαράμ. Αλλά πιστεύω παρόλα αυτά υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Μια μικρή φλόγα ελπίδα στην Ιγυρία. Άλλαξε η κυβέρνηση, άλλαξε το δημοκρατικό καθεστώ με ειρηνικό τρόπο. Δεν είναι αυτονόητο αυτό στην Αφρική και ο νέο πρόεδρο υπέβαλε ένα πρόγραμμα πολλά υποσχόμενο και μεταξύ άλλων υπόσχεται και την καταπολέμηση της διαφθοράς, την προστασία των γυναικών και την χρήση της στρατού κατά της Μπόκο Ελπίζουμε, ελπίζουμε να πετύχει η εφαρμογή του προγράμματος αυτού και νομίζω ότι θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να υποστηρίξουμε και την περιοχή και την κυβέρνηση προκειμένου να σταθεί με επιτυχία το νέο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρος. Τελευταίος εισηγητής. Φίσας Αϊσέλα. Ευχαριστώ σε επικεφαλή τη Επιτροπή Εκλογική Παρατήρηση στην Ιγυρία. Πήγα τέσσερι φορέ φέτο και θα ξαναπάω και τη Δευτέρα για να ε, υποβάλω στην κυβέρνηση την τελική μου έκθεση. Είναι πραγματικά ε, τρομακτική η κατάσταση στη χώρα λόγω των επιθέσεων ε, τη τρομοκρατική ομάδα Μπόκο Χαράμα. άκρο επώδυνε η κατάσταση των χιλιάδων κοριτσιών που έπεσαν θύμα βιασμού, έχουν εξισλαμιστεί, αναγκάζονται να παντρευτούν και πολλές φορές χρησιμοποιούνται ως καμικάζι αυτοκτονίας, αλλιώς ε, θα τις θάψουν ζωντανές. Και πολλές χιλιάδες ε, άνθρωποι έχουν καταλήψει τα σπίτια τους και περιφέρονται εκτοπισμένοι. Δεν πρέπει να ε, μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα μπροστά σε αυτές τις φρικαλαιότητες. Πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις και δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει να στηρίξουμε και την νέα κυβέρνηση αλλά και την Ένωση των Αφρικανικών χωρών αυτό το τη συμμαχία που επιτέλους έχουν οργανώσει κατά της Μποκοχαράμ. Ευχαριστώ. Σάντσες, ε, επόμενο, επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ πολύ η Νιγηρία είναι η πολυπληθέστερη από τι πιο πλούσιε και μεγαλύτερε οικονομίε τη Υπήρου. Με πολύ ορυκτό πλούτο, πετρέλαιο. Όμω πάνω από 70 εκατομμύρια ε, κάτοικοι τη χώρα ζουν κάτω από το όριο τη φτώχεια. Ανισότητα, ε, ε, απόγνωση είναι το καλύτερο, το πιο πρόσφορο έδαφο για την ανάπτυξη τη βία. Σίγουρα πρέπει να παρασχεθεί ανθρωπιστική βοήθεια. Τα αίτια όμω πρέπει να τα αναστήσουμε και σε εξωτερικέ δικέ μα πολιτικέ, όπω είναι η εμπορική πολιτική που φτωχαίνουν Αφρική. Τα παιδιά είναι τα βασικά, τα κύρια θύματα της βίας. Ε, απάγονται, ε, στρατολογούνται και υπό, ε, υπόκεινται σε σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση από την Πόκο Χαράμ. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς. Εάν με την εμπορική μας πολιτική συνεχίσουμε να φτωχαίνουμε την Αφρική και δεν κάνουμε τίποτε για να προωθήσουμε ένα δίκαιο φορολογικό και ένα διανεμητικό σύστημα σε όλο τον κόσμο, τότε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα φαινόμενα και δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το προσωπικό πρόσωπό ε, Αυτό θα πει Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την ομιλία σας, σας ευχαριστώ και για το έργο των ε, εισηγητών τώρα από τις ομάδες. Θα ακούσουμε τους ομιλητές. Πρώτος ομιλητής από το ΕΛΚ, ο κύριος Κέλλη. Έχει το λόγο. Κύριε Κέλλη, έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό μάλλον. Ε, Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Ήμουν σε τριμερή διάλογο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό και θα πρέπει να το εξετάσουμε υπό το πρίσμα των συζητήσεων που διεξαγάγονται στο Κοινοβούλιο και που έγιναν και με την καγκελάριο κυρία Μέρκελ, τον πρόεδρο Ολάντ οι οποίοι επισήμεναν ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στην Αφρική να δώσουμε υποστήριξη σε σημαντικά συντήματα όπως η αλλαγή του κλίματος και σε ό,τι αφορά την δημιουργία καλύτερων όρων διαβίωση για αυτού που ζουν εκεί. Κοιτώντα λοιπόν τι συμβαίνει στην Ιγυρία, βλέπουμε πόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστούν ε, ομάδε οργανώσει όπω η Μπόκο Χαράμ και η τρομοκρατία που πλήττει κυρίω ε, του νέου, νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που στράφεται κατά των σχολείων των ίδιων. Είναι σαφές λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη και με όλους τους άλλους φορείς για να δημιουργηθούν καλύτεροι όροι διαβίωση. Και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Κέλλη λέει η Πρόεδρος. Μπλε κάρτα έχετε. Την αποδέχεστε. Από τον κύριο Ρούμπιχ. Ναι, κύριε Ρούμπιχ, έχετε λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον ε, συνάδελφο Κέλλη τι γίνεται με το έργο για την εκπαίδευση. Υπάρχει δυνατότητα να ε, δοθεί ε, εργασία κατάρτισης, παιδείας, προκειμένου να τεθούν οι κατάλληλοι όροι και συνθήκες. My colleague, Mr. Rubik, is absolutely correct. Απόλυτο δίκαιο, συνάδελφος Ρουμπίχ. Απόλυτο δίκαιο άλλο να καταπολεμήσουμε την Μποκοχαράμ και άλλο να δημιουργήσουμε μια ανατροπία, μια κουλτούρα σεβασμού και αναγνώρισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ε, ατόμων. Και μόνο με ένα σύστημα σωστό εκπαίδευσης ε, και παιδείας μπορεί να συμβεί αυτό. Άρα λοιπόν ε, το να δημιουργούμε σχολεία και άλλο αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ιγυρία. Και αν δεν υπάρχει πραγματικά ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν θα υπάρξει ποτέ πραγματική πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ρουμπίχ. Ευχαριστώ, λέει και η πρόεδρο. Και πάρω να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλενσιανό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα συνηθίζουμε τις ε, τραγωδίες ε, που μας ε, περιτριγυρίζουν, που μας περιβάλλουν και πολλά πρωινά, πολλά απογεύματα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, για εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια που δέχονται βάρτατες επιθέσεις και δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να τους στερείς την παιδεία, την εκπαίδευση τους δεν είναι τίποτα χειρότερο για τα παιδιά από το να τους στερείς κανείς την εκπαίδευσή τους και μπορεί να συνηθίσουμε σιγά σιγά αυτά τα νούμερα. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι οι δωρητές, ε, ε, εμείς ε, που έχουμε δεσμευθεί να παρέχουμε κάποια κονδύλια ώστε να μπορεί να γίνει πραγματικότητα εκπαίδευση αυτών των παιδιών και για να υπάρξει και αποτελεσματική καταπολέμηση της Μπόκο Χαράμ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Δηλαδή τρία ευρώ δεσμεύουμε ότι θα δώσουμε, δεσμεύουμε ότι θα δώσουμε και τα δύο τα χρωστάμε τελικά. Πρέπει όμως ε, και τα κράτη-μέλη να καταλάβουν ότι πρέπει να αναλάβουν ε, τις ευθύνες τους ε, και να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για να πάψουν αυτές οι βαρβαρότητες στην Νιγηρία. Και απευθύνουμε και στον πρόεδρο τον καινούριο της χώρας. Ευχαριστώ. Μπέλντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην παράγραφο 11 της, του κοινού ψηφίσματος αναφέρεται μία φράση η οποία με άγγιξε. Παραθέτω εκφράσουμε την απόλυτη συμπόνια για τα παιδιά και τις γυναίκες που υπόκειται την τυφλή, τη τυφλή βία της Μπόκο Χαράμ και επέζησαν. Και έχω υπόψη μου τον Χάσαν Μπέτρους, ε, τεσσάρων ετών από την Ιγυρία, από την Βόρεια Ιγυρία, το Δεκέμβριο Βγήκε με ένα βίβλο από την εκκλησία και οι εξτρεμιστές της Μποκοχαράμ το σταμάτησαν, του πήραν τη βίβλο από το χέρι και την πέταξαν σε ένα σε μια φωτιά. Ο Χασάν προσπάθησε να βγάλει τη βίβλο με ένα ξυλαράκι από την πυρκαγιά, από τη φωτιά. Και τον πέταξαν μέσα στην φωτιά τα μέλη της Χαράμ. Ευτυχώς επέζησε ο Χασάν λοιπόν και όλα τα θύματα της Μπόκο Χαράμ ζητούν ε, παραπάνω από συμπόνια. Ζητούν διεθνή προστασία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και συμφωνούμε από αυτόν, λέει η Πρόεδρο. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Βάτμαντσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Συνάδελφοι, πιστεύω ότι όλοι το είπαν σήμερα ότι πρέπει να μιλήσουμε για το θέμα τη Νιγηρία. Πάνω από ένα εκατομμύριο παιδιά έχουν φύγει και διώκονται. Τα πιο πολλά κάτω των πέντε χρονών και οι που δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο γιατί απειλείται η ζωή τους. Η Μπόκο Χαράμ, ξέρετε συνάδελφοι, φοβάται τους ανθρώπους που έχουν άποψη. Τόσο δειλή είναι και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την Μπόκο Χαράμ. Θα πρέπει φυσικά να προσέξουμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε από τον νέο πρόεδρο να κάνει έρευνα για την παραβίαση δικαιωμάτων από τα πρώην μέλη του στρατού. Και θα ήθελα να πω και δύο λόγια για τις μαζικές βιασμούς ε, γυναικών. Θα πρέπει να κάνουμε μία έκκληση. Θα πρέπει να τους επιτρέψουμε να κάνουν εξτρώσεις, αμβλώσεις σε περίπτωση που μετά τα εγκλήματα αυτά μένουν και έγκυες από πάνω. Σας ευχαριστώ και διακόπτη πρόεδρο. Σας Ευχαριστώ. Ε, κύριε Σομπερμαϊερ, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Εδώ και χρόνια ακούμε τις εκκλήσεις ε, για την καταπολέμηση, την πιο έντονη καταπολέμηση της Μποκο Χαράμ. Συμπεριλαμβάνονται τέτοια θέματα λοιπόν στη ημερήσια διάταξη και το καλοκαίρι είδαμε τι έγινε με τα παιδιά στρατιώτες και με την ε, καταστροφή χριστιανικών χωριών στην ε, Βόρεια Νιγηρία έχουμε 1,2 εκατομμύρια παιδιά που έχουν φύγει από τα σπίτια του και σύμφωνα με τη UNICEF και τα στοιχεία της το ίμιση είναι κάτω των 5 ετών. Αν η Ευρώπη λοιπόν ε, θέλει να εντατικοποιήσει και αν, δεν, ε, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συστηματοποιήσει την καταπολέμηση της Μποκοχάραμ να μην ε, μείνουμε έκπληκτοι στο επόμενο τσουνάμι προσφύγων που θα καταφτάσει στην Ευρώπη, αγαπητοί συνοδελφοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Ένα λεπτό, κύριο Σέτμαν. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η σύραξη στην Ιγυρία έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 20.000 ανθρώπους, ενώ εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί. Και δεδομένη της κοινωνικής δομής της Νιγηρίας, όπου το 40% των ανθρώπων είναι κάτω το... είναι πολύ νέοι, τα περισσότερα θύματα είναι παιδιά. Ε, ε, είναι θύματα βίας, αλλά και θύματα της έλλειψης παιδείας ή ε, κοινωνική περίθαλψης. Δεν έχουν κανονική παιδική ηλικία. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια καθολική προσπάθεια και βελτίωση της κατάστασης στη χώρα, ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά όχι μόνο. Και Είμαι ευχαριστημένος που η Κομισιόν έχει δώσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ πρόσφατα Πάντως πρέπει να γίνουν και περισσότερα ακόμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ συνάδελφε. Ο κύριος Γιούζα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τόσα συμβαίνουν στην Ιγυρία είναι πράξεις ε, τεράστια και απίστευτης βαρβαρότητας. Εγώ είμαι υπέρ του να λάβει, κάνει κάποια βήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να απαλύνει την τραγική κατάσταση στην οποία ζουν οι άνθρωποι της Νιγηρίας. Παιδιά, γυναίκες ε, και όλα τα θύματα. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι αρχές της χώρας θα πιεστούν και θα ενεργήσουν. Θα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για το γεγονός ότι η κοινωνία μισεί το χριστιανισμό ε, ε, και θα πρέπει αυτό να το αναφέρουμε και στο ψήφισμά μας ξεκάθαρα. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλντ έχει το λόγο τώρα. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι, μισό εκατομμύριο παιδιά έχουν ε, αρπαγεί από τα σπίτια τους και έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους εδώ και έξι χρόνια που η Μπόκο Χαράμα ε, τρομοκρατεί τον κόσμο μέσα και γύρω από την Ιγυρία. Θα πρέπει να είμαστε κατά της ε, δουλείας των καταναγκαστικών γάμων το, οποιασδήποτε μορφής βίας κατά των παιδιών. Ε, η, καρδιά μας θα πρέπει να, και το μυαλό μας θα πρέπει να είναι στα θύματα και στις οικογένειες. Θα πρέπει τουλάχιστον να θυμηθούμε τις μαθήτρες του ΣΥΜΠΟΚ που έχουν απαχθεί πριν από 1,5 χρόνια, 1,5 χρόνο και χιλιάδες παιδιά ε, που έχουν απαχθεί στην Ιγυρία. Δεν θα πρέπει να τα ξεχάσουμε αυτά τα παιδιά, να γνωρίζουν ότι δεν είναι μόνο τους. Πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα, να κινητοποιηθεί η στήριξη στην Ευρώπη, ώστε να ενώσουμε τις δυνάμεις με την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, ώστε να στηριχθεί η κυβέρνηση της Νιγηρίας και η Αφρικανική Ένωση για να μπορέσει να προστατέψει τα παιδιά, να ερευνήσει αυτά τα εγκλήματα και να θέσει τέλος στην ατιμορρησία. Τα παιδιά θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στις βασικές βασικές ανάγκες, νερό, φαΐ, κατάλημα, ε, ε, υγεία και σχολείο. Εμείς θα συνεχίσουμε να κρατούμε στη μερίσια διάταξη τη μοίρα των παιδιών αυτών στην Ιγυρία όσο χρειαστεί. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση με τους μεμονωμένους ομιλητές και Έχω οκτώ βουλευτές που έχουν ζητήσει το λόγο στη διαδικασία Catch the Eye. Θα ακολουθήσω τη σειρά με την οποία ζήτησαν το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ με τα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ του συντάκτε αυτού του ψηφίσματο και όλου όσου πήραν το λόγο σήμερα και καταδίκασαν τη βία που πει στην Ιγυρία. Τα νούμερα τα είπαμε. Δύο εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι άνθρωποι, χιλιάδε δολοφονίες ε, παιδιών, γυναικών, πάνω από 10 εκατομμύρια παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο στην Νιγηρία. Είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ε, κατακεφαλήν σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, ε, πρέπει αυτό να το ζητήσουμε. Δεν πρέπει να το υποτιμάμε ως στοιχείο επειδή δεν μας αφορά άμεσα. αντίθετα με τα προβλήματα της Μέσης Ανατολής. Εγώ πιστεύω πως θα πρέπει η Κομισιόν να δραστηριοποιηθεί ακόμη περισσότερο, να ηγηθεί στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας <clears throat> στα παιδιά και στις γυναίκες σε αυτή την περιοχή. Είναι απαραίτητο τα χρήματα που υποσχέθηκαν οι δωρητές να δοθούν και συντονισμό να γίνει με τον νέο πρόεδρο της Νιγηρίας. Ο κύριος Γιούρεκ είναι ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Μποκοχαράμ θεωρούσαμε πριν από κάποια χρόνια ότι θα υποχωρήσει και ότι θα ακούμε όλο και λιγότερα ε, για τη δραματική κατάσταση των ε, παιδιών μετά τη δράση της ε, κυβέρνησης. Δυστυχώς όμως εξακολουθεί να δράει ε, Μπόκο Χαράμ διότι η κυβέρνηση έρχεται στα λόγια και δεν ε, αναλαμβάνει ε, δράση. Αυτά που συμβαίνουν Αφρική, Νότος, περιοχή μεγάλων λιμνών, Κεντρική Αφρική. Πρόκειται για μία από τις πιο σοβαρές γεωπολιτικές τραγωδίες τόσο στην Ήπειρο αυτή όσο και στον κόσμο συνολικά. Είναι μια ανθρωπιστική τραγωδία οι κάτοικοι των Αφρικανικών χωρών αλλά και η γυριανή ε, κυβέρνηση δεν ε, ε, μπορεί να αρκείται πλέον στο να, να δίνουμε όλο και περισσότερα ψηφίσματα στη δημοσιότητα. Χρειάζεται δράση. Ο κ. Αφρουντσούλικα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και ε, αστάθεια λόγω της, ε, των ε, συγκρούσεων μεταξύ Μπόκο Χαράμ, στρατού και άλλων ομάδων. 500.000 παιδιά εκτοπισθέντα ε, στη βόρειο-ανατολική Νιγηρία και στο Νίγηρα και συνολικά 1,4 εκατομμύρια παιδιά εκτοπισθέντα τα οποία κινδυνεύουν να μπουν σε αυτό τον φαύλο κύκλο βίας για πάντα. Τα εκμεταλλεύονται, τα στρατολογούν. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα δώσει χρήματα για την ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Υπάρχει όμως ένα κενό χρηματοδότησης και υπάρχει και ε, για τις ε, επιχειρήσεις της UNICEF ένα κενό μεταξύ των πιστώσεων πληρωμών και των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποκαταστήσουμε τη σταθερότητα στη χώρα, να αντιμετωπίσουμε την πόκο χαράμ αλλά και τα βαθύτερα αίτια τη λαβομετανάστευσης και της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η τρομοκρατία σήμερα αποτελεί το πιο μεγάλο ζήτημα στον κόσμο. Απειλεί όλους τους ε, πολίτες, ανεξάρτητα α, της καταγωγής τους και του τόπου γέννησης τους. Και η Μπόκο Χαράμ αποτελεί μαρτυρία αυτού. Αυτή η τρομοκρατική λοιπόν οργάνωση αποτελεί αυξανόμενη απειλή για την ασφάλεια της Βορειοαφρικής και της Νιγηρίας. Συνεχίζουν τις απαγωγές, τις ε, επιθέσεις αυτοκτονίας και επεκτείνουν και τι δραστηριότητε του οι γειτονικέ χώρε. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να υποστηρίξω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη δήλωση που έκανα, που καλεί τη διεθνή κοινότητα για μεγαλύτερου πόρου και ανθρωπιστική βοήθεια. Από κοινού λοιπόν με τη διεθνή κοινότητα πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον ε, νέο εκλεκτέντα πρόεδρο τη ε, Νιγηρία και να πάρει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ε, πολιτών της Νιγηρίας, ιδιαίτερα τους γυναίκες και τα παιδιά και να παρέχει προστασία για τα θύματα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και δώσω τον λόγο στην κυρία Λόχμπιλερ τώρα. Αν δεν είναι εδώ η κυρία Λόχμπιλερ. Καστάλτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν δούμε τα νέα που μας στάνουν από την Αιγυρία, δυστυχώς ε, διαβάζουμε ένα πολεμικό ανακοινωθέν. Ε, γυναίκες, παιδιά, κοριτσάκια 5 με 14 ετών χρησιμοποιούνται με σχρό τρόπο για επιθέσεις καμικάζι. Ο ΙΕ μέσω της UNICEF είπε ότι χρειάζονται ε, πολλά χρήματα, αλλά μόνο το 32% αυτών έχουν φτάσει για να αντιμετωπιστεί αυτή η επίγουσα ανάγκη. Οι διεθνεί δωρητέ ε, θα πρέπει να κάνουν κάτι παραπάνω από το να δίνουν χρήματα. Να κάνουν περισσότερα για να προστατευτούν οι άμαχοι και για να μπορέσουν αυτά τα κοριτσάκια που έχουν βιαστεί να ε, λάβουν την απαραίτητη υγειονομική περίθαψη και την άμβλωση αν χρειάζεται. Πρέπει να έχουμε διορατικέ και βιώσιμε πολιτικέ και να επανέλθουμε στην πηγή του θέματο τη τρομοκρατία δημοκρατία, σε φτώχεια, ανεπαρκής ε, διακυβέρνηση. Ε, δεν θα λύσουμε ποτέ το πρόβλημα αν δεν επανέλθουμε στι ρίζε λοιπόν του προβλήματο, ούτε στην Ιγυρία ούτε κι αλλού. Να, να αλλάξουμε και να καλύψουμε τι κρίσει αλλάζοντα τη δική μα συμπεριφορά. Σα ευχαριστώ. Πετήρ. Σας ευχαριστώ και καταδικάζω την ε, Χαράμ και τις δράσεις που προκαλούν τέτοια πόνο και τέτοια α, βία στα παιδιά και στις, ε, στα κορίτσια, όχι μόνο στην Ιγυρία, αλλά και στον Ήγυρα, στο Τσάτ, στις γειτονικέ χώρες. Είναι απαράδεκτο να μην μπορούν τα παιδιά να πάνε στο σχολείο και να χάνουν την αθότητα της παιδικής τους ηλικία. Να τα βγάζουν από τους κόλπους της οικογένειάς τους και θα ήθελα να πω ότι αυτή η τρομοκρατική οργάνωση ε, έχει βάλει στο στόχαστρο τους χριστιανούς έχουν χαθεί 10.000 ζωές τα τελευταία χρόνια. 250.000 άτομα είναι εκτοπισμένα. Οι δολοφονίες λοιπόν της ε, Μποκοχαράμ αποτελούν εγκλήματα και αυτό είναι απαράδεκτο και καλό όλους τους φορείς να καταδικάσουν τις ε, εγκλήματα αυτά. Θα πρέπει να είναι σαφής η αντίδρασή μας, να σταματήσουμε τις οικονομικές ροές προς την Μπόκο και να ενισχύσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια προς τα παιδιά τα οποία φεύγουν από τις περιοχές αυτές που είναι... Κυρίες Μαμικιάς. Πρόεδρε, η Νιγηρία είναι μια πλούσια χώρα, με πλούτο παραγωγικές πηγές, με πετρέλαιο, με τεράστια έσοδα. Και όμως ο πληθυσμός στην Νιγηρία ζει μέσα στη φτώχεια και βρίσκεται αντιμέτωπος με την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έτσι η υπανάπτυξη η έλλειψη δημοκρατίας και η διαφθορά αποτελούν λίπασμα για την τρομοκρατία και την ανάπτυξη της μπόκο χαράμ της οργάνωσης αυτής των τζιχαντιστών που συνεργάζεται στενά με τον ίσις. η μπόκο χαράμ λοιπόν αναπτύσσεται συνεχώς ασκεί τρομοκρατία είναι υπεύθυνη για δολοφονίες για βομβιστικές ενέργειες για απαγωγές παιδιών για βιασμούς. από το 2009 εκατομμύρια παιδιά έχουν εγκαταλείψει τις αιστείες τους για να σωθούν. για να ιτηθεί η μπόκο χαράμ πρέπει να χτυπηθεί η φτώχεια πρέπει να χτυπηθούν τα αίτια που δημιουργούν την τρομοκρατία πρέπει τα τεράστια έσοδα από το πετρέλαιο στην Ιγυρία να πάνε υπέρ του ίδιου του λαού της νιγηρίας και όχι στις τσέπες των πολυεθνικών. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εδώ ολοκληρώθηκε η διαδικασία Catch με τον τελευταίο μιλητή. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου ε, για τα θύματα και της επίσης προηγουμενής εβδομάδα. Ε, πρέπει να στηρίξουμε την υγεία και την κυβέρνηση της χώρας στον αγώνα που δεν είναι κατά της Μποκοχαράμα που έχει τόσα θύματα. Ο πρόεδρος Μπουχάρη ε, πρέπει να προσκληθεί στο κοινοβούλιο, ε, θα έρθει του χρόνου. Σίγουρα χρειάζεται η ανθρωπιστική βοήθεια, αλλά χρειάζεται στήριξη και η Νιγηριανή κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα βαθιά αίτια που είναι η ακραία φτώχεια, κοινωνικέ ανισότητε, ε, η δημική διαφθορά. Είναι απαράδεκτο μια τόσο πλούσια χώρα να έχει τα δύο του πληθυσμού της να ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κάτι που αποτελεί πρόσφορο έδαφος ε, για τη ριζοσπαστικοποίηση. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ε, και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου πρέπει να καταπολεμηθεί διαφθόρα. Ευχαριστώ. Τώρα ολοκληρώθηκε λοιπόν η διαδικασία κάτσε διάλειο ο πρόεδρος, ο κύριος Τηλιανίδης, ο επίτροπος απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνόλοι, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την δυνατότητα να σχολιάσω την ανθρωπιστική κατάσταση στην Βορειοανατολική Νιγηρία και ιδίως την κατάσταση των παιδιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και την πολύ πλούσια αυτή συζήτηση. Ήμουν ε, στην περιοχή πριν από δύο-τρεις μήνες, επισκέφθηκα ε, τις ε, Περιοχέ που είναι πολύ κοντά στην περιοχή που ελέγχει Μπόκο Χαράμ και είναι σαφές ε, ότι η βία ε, της Μπόκο Χαράμ ε, παραμένει άκρο ανησυχητική και δυστυχώς δεν έχουμε κάποιες, κάποιες ενδείξεις για βελτίωση στο άμεσο μέλλον. Έχουν βέβαια από τη νέα Νιγηριανή κυβέρνηση επιτευχθεί κάποια βήματα πρόοδου κατά της υποκοχάρμης συνεργασία και με τις ε, γειτονικέ χώρες. Όμως έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση επιθέσεις ε, της Μποκοχάρμ. Και αυτό ε, και περισσότερη οδύνη πόνο και αστάθεια προκαλεί, αλλά βλέπουμε να χρησιμοποιούνται τα παιδιά ως όπλα για την για τις επιθέσεις αυτοκτονίας. Πρόκειται για κάτι απαράδεκτο και πραγματικά πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι, προσιλωμένοι στο στόχο να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο. Πρόκειται για μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο. Ο αριθμό των εσωτερικά εκτοπιστέντων ατόμων στην Ευανατολική Νιγηρία έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Συνολικά, ε, στην περιοχή των Λιμνών και στο Τσάντ, 700.000 παιδιά κατέληψαν τη αιστείας του και τα περισσότερα από αυτά μένουν, φιλοξενούνται όχι σε επίσημους καταβλισμούς και οι ανάγκες τους ό,τι αφορά ε, τροφή, στέγαση, υγεία, παιδεία δεν καλύπτονται τις περισσότερες φορές ε, επειδή είναι πολύ ευάλωτα γίνονται και εύκολα θύματα ε, κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Εμείς παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση μαζί με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ε, και τον ΟΗΕ βοηθούμε με διάφορα μέσα την Ιγυρία καταρχάς με την ανθρωπιστική βοήθεια, στην ε, υγειονομική περίθαλψη, επιστηστική ασφάλεια, ε, διατροφή, προστασία, ε, κατάλήματα και εστιάζουμε ειδικά στα παιδιά στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας. Είμαστε ο πρώτος δωρητής στην Ιγυρία από τότε που ξέσπασε η κρίση της Μποκοχαρά. Έχουμε κινητοποιήσει 20,5 εκατομμύρια μόνο για το τρέχον έτος και 32,5 εκατομμύρια για την περιοχή των Λιμνών και του Τσάντ. Θα παράσχουμε επίσης υποστήριξη και στην πολυεθνική κοινή ομάδα δράσης που έχουν συγκροτήσει, που συγκροτούν μάλλον ε, οι ε, χώρες ε, της περιοχής 50 εκατομμύρια περίπου έχουμε ε, υπολογίσει ως ποσό θα χρειαστεί, αλλά για τη δέσμευση των κονδυλίων απαιτείται η ε, υλοποίηση κάποιων προϋποθέσεων και θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες αν θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Επίσης χρηματοδοτούνται ειδικά τρομοκρατικά προγράμματα που καταπολεμούν την ε, ριζοσπαστικοποίηση και έχουμε μέτρα ε, για το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις αθλητικές επιχειρήσεις. Με την, ε, μεταξύ άλλων, ε, την βελτίωση της αντίδρασης του δικαστικού συστήματος, στη δρομοκρατία, τη βελτίωση των επικοινών κτλ. Στο πλαίσιο του ΕΤΑ ε, προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα βαθύτερα αίτια της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας, πάλι εδώ ε, κυρίως έχοντας υπόψη στα παιδιά. Υπάρχει ένα σχέδιο ε, παιδικής προστασίας ό,τι αφορά και τη δικαιοσύνη ανηλίκων, την υγεία, ψυχοκοινωνική μέρημνα για τα παιδιά και τους νέους που ζουν σε εμπόλεμε περιοχές και γενικότερα προσπάθεια ανοικοδόμηση τη Βορειοανατολική Νιγηρία. Η Νιγηρία επίσης είναι μια χώρα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά ε, την πρωτοβουλία μας για τα παιδιά σε εμπόλεμέ. περιοχές. Η χώρα ε, περιλαμβάνεται ε, στον κατάλληλο στην έκθεση του ΟΗΕ για τις για το θέμα αυτό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση ε, και ε, να περιορίσουμε ε, τα βάσανα των παιδιών λόγω της βίας της Μποκοχάραμ. Δυστυχώς όμως η εθνική κυβέρνηση είναι αυτή που πρέπει να κάνει τα δέοντα. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με την κοινότητα των πολιτών και με τα Ηνωμένα Έθνη και με τους ανθρωπιστικούς φορείς επιτόπου θα συνεισφέρουμε όσο μπορούμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε, για τα καταληκτικά σας σχόλια και λάβαμε επτά σχέδια ψηφίσματος. Τώρα, λοιπόν, ολοκληρώνεται η συζήτηση αυτή.